περιφέρεια είναι μια περιφέρεια συνύπαρξης της φύσης και του ανθρώπου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. Σας ευχαριστούμε. Περνάμε τώρα αγαπητοί συνάδελφοι στο επόμενο σημείο που είναι η έκθεση της Σιλβάνα Δράπτη Καθολική Υπηρεσία και αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης 112. Δίνω το λόγο στην εισηγήτρια, στην κυρία Σιλβάνα Ράπτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχω πόσα λεπτά. Έχω πόσα λεπτά. Όσα και να έχω, έχω χάσει λίγο χρόνο από τη μετάφραση. Ξεκινώ και σταματάτε εσείς την... Sorry, sorry, you have, you, have, you have, minutes. Τέσσερα λεπτά. Ε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η έκθεση την οποία ε, πραγματεύομαι έχει θέμα τον πανευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 και την καθολική υπηρεσία. Ο αριθμός 112 είναι πάρα πολύ χρήσιμος, αλλά όσο χρήσιμος είναι τόσο λίγο γνωστός είναι με βάση τα στοιχεία που έχουμε από το ευρωβαρόμετρο το φεβρουάριο του 2011 βλέπουμε ότι μόνο το 26% των ευρωπαίων πολιτών μπορούν να συνδέσουν τον αριθμό 112 με την χρήση που μπορεί να έχει για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. ο στόχος μας πρέπει να είναι ως το δύο το ποσοστό των πολιτών που θα μπορούν να συνδέσουν τον αριθμό 112 με την κλίση έκτακτης ανάγκης να φτάσει το 80%. Ένας στόχος φιλόδοξος, ο οποίος για να γίνει πραγματικότητα χρειάζεται να γίνουν προηγουμένως κάποια άλλα πράγματα. Τα πράγματα αυτά είναι κατά τη γνώμη μου τρία. Το πρώτο είναι η ενημέρωση. Η ενημέρωση μπορεί να περάσει μέσα από τα σχολεία και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως επίσης μέσα από τους σταθμούς εισόδου των τουριστών σε κάθε πόλη πράγμα που σημαίνει ότι το 112 πρέπει να διαφημίζεται στα λιμάνια στα αεροδρόμια στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. το δεύτερο σημείο είναι το θέμα της καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των 27 χωρών μελών της ευρωπαϊκής ένωσης. καταλαβαίνουμε όλοι πόση σημασία έχει ένας ευρωπαίος πολίτης ιδιαίτερα τώρα που είναι καλοκαίρι που ξεκινάει η περίοδος των διακοπών να μπορεί να έχει την ασφάλεια να ξέρει ότι καλώντας το 112 θα λυθεί το πρόβλημά του σε οποιαδήποτε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης και αν βρίσκεται σε οποιαδήποτε γλώσσα και αν απευθυνθεί στο τηλέφωνο. το βασικότερο όμως σημείο απ' όλα είναι η εντόπιση της θέσης του καλούντος να μπορούμε κατευθείαν να εντοπίσουμε πού βρίσκεται αυτός που έχει πρόβλημα και να τον βοηθήσουμε. εδώ έρχεται η τεχνολογία. εδώ η τεχνολογία παίζει καθοριστικό ρόλο και εδώ κάπου έρχεται και εμπλέκεται και το ζήτημα της καθολικής υπηρεσίας. να ξέρουμε γιατί μιλάμε και να ξέρουν και οι πολίτες που μας ακούν. η καθολική υπηρεσία το ξέρουμε όλοι ότι είναι μια στοιχειώδης δέσμη υπηρεσιών καθορισμένης ε, ποιότητας που να μπορεί να παρασχεθεί σε προσιτή τιμή και χωρίς να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. αυτό είναι μια έννοια που εμπεριέχεται στην οδηγία που είχε εκπονηθεί το 2002, μια οδηγία η οποία αναθεωρήθηκε το 2008 και που μόλις το Μάιο τελείωσε η περίοδος που έχουν τα κράτη μέλη για να ενσωματώσουν την οδηγία αυτή μέσα στο δίκαιό τους. κατά συνέπεια τώρα μόλις αρχίζουμε να έχουμε την περίοδο αξιολόγησης πράγμα που θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό πριν προχωρήσουμε σε ένα επόμενο στάδιο. και αυτό το λέω διότι την κουβέντα αυτή την κάνουμε σε μια περίοδο που είναι εξαιρετικά κρίσιμη για τα οικονομικά της ευρωπαϊκής ένωσης και για τα οικονομικά των χωρών μελών. Ε, θεωρώ απαραίτητο να τονίσω ότι η καθολική υπηρεσία κατά τη γνώμη μου δεν είναι ούτε η μοναδική αλλά ούτε και η βασική όθηση για να, ε, πετύχουμε τον στόχο της ευρυζωνικότητας για όλους. και αυτό γιατί απαιτείται πολύ υψηλό επενδυτικό κόστος χωρίς κατά ανάγκη να έχουμε σημαντικά βελτιωμένες υπηρεσίες στους καταναλωτές. Ε, θέλω δε στο σημείο αυτό να πω και δύο αριθμούς που έχουν τη σημασία τους. Σαφώς και υποστηρίζω την ψηφιακή ατζέντα και τους στόχους της, αλλά όταν βλέπουμε ότι ακόμα και εκεί που είναι στο 100% διατιθέμενη ευρυζωνικότητα γίνεται χρήση μόνο στο 50%, αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Ε, νομίζω ολοκληρώνοντας κύριε πρόεδρε ότι η εισαγωγή της υποχρέωσης της ευρυζωνικότητας στην καθολική υπηρεσία θα πρέπει να ακολουθηθεί από κάποια συγκεκριμένα μέτρα και παροχή κινήτρων στον ιδιωτικό τομέα με χρηματοδότηση και από εθνικούς και από κοινοτικούς πόρους. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Έχουμε διάφορους ομιλητρίες που έχουν ζητήσει το λόγο. Η κυρία Μπασέσκου είναι η πρώτη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ενιαία αγορά θα πρέπει να εξασφαλίζει πρόσβαση για όλους τους πολίτες Νομίζω ότι με αυτή την έκθεση προσφέρονται πάρα πολλές λύσεις για αυτό το πρόβλημα. Ε, με, αυτή, με αυτόν τον τρόπο θα προαγάγουμε την κοινωνική συνοχή καθώς και τις διασυνοριακές επενδύσεις. Η σωστή εφαρμογή της οδηγίας για τις καθολικές υπηρεσίες είναι το κλειδί για μια εύρυθμη εσωτερική αγορά. Ο αριθμός κλήσης 112 είναι μια από τις επιτυχημένες ιστορίες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να συνεχίσουμε την εκστρατεία ενημέρωσης ε, των πολιτών και καλωσορίζω το ότι οι αρμόδιες ε, για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ανάγκες αρχές ε, είναι ενημερωμένες και προωθούν αυτόν τον αριθμό επίσης. Ε, καλό θα ήταν ε, να σημειωθεί η πρόοδος για τον εντοπισμό του καλούντος, γιατί κάθε λεπτό μετράει. Σας ευχαριστούμε, Μάλικομ Χάρμπορ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε ως πρόεδρος της Επιτροπής και ως κοιόδης εισηγητής ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ράπτη. Εκπώνησε μια εξαιρετικά ισορροπημένη και λίαν σημαντική έκθεση ε, και συμβάλλει στην αναθεώρηση που έχει ήδη ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλωσορίζω την παρουσία της κυρίας Μάλμστρομ. Ε, ξέρω ότι ιδιαίτερα στην ε, Σουηδία, όπως και άλλες χώρες, καταβάλλουν τις προσπάθειες για την πρόθεση της ευρυζωνικής σύνδεσης. Ε, η κυρία Ράπτη ε, μας λέει ότι είναι παροχημένες οι διατάξει για τις καθολικές υπηρεσίες, το ξέρω κι εγώ ίδιος, ε, γιατί από το 99 ασχολούμαι με αυτό το ζήτημα και τότε τα κινητά ήταν νεογνά. Τώρα ε, έχουμε βρεθεί σε μια θέση όπου ε, κατά μέσο όρο όλοι μας έχουμε πάνω από ένα κινητά. Οπότε αυτή η ιδέα της καθολικής υπηρεσίας ε, θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί, να επαναδιαμορφωθεί. Τώρα με την ευρυζωνική σύνδεση έχουμε πάρα πολλά προγράμματα βάσει των οποίων οι κυβερνητικές αρχές έχουν αναλάβει δέσμευση για τις καθολικές υπηρεσίες. Να μεριμνήσουμε ώστε να εφαρμοστούν τα προγράμματα, αλλά να μεριμνήσουμε επίσης ο χρόνος σας κύριε Χάρμπορ να μεριμνήσουμε, έλεγα, ώστε οι άνθρωποι με αναπηρίες να έχουν επίσης πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες ε, και οι κείμενοι, οι νομικοί όροι πρέπει να ενισχυθούν για να συμβεί αυτό. Σας ευχαριστώ, κύριε Χάρμπορ. Η κυρία Ρουιτόβου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που ακούσαμε από τους συναδέλφους. Ε, το πρόβλημα της, ε, του αριθμού 112 είναι ότι δεν είναι γνωστό από τους πολίτες. Άρα θα πρέπει να ε, συνεχίσουμε την εκστρατεία ενημέρωσης. Επίσης, στο κολάριο εντοπισμού πρέπει να προωθηθεί η διάταξη περιοντοπισμού του καλόντος ε, κατόπιν θα προσέθετα ότι χρειαζόμαστε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Υποστηρίζω επίσης ε, τις διατάξεις που μας προτείνει η συγγήτρια για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ε, και καλό την Επίτροπο να προωθήσει το θέμα της ε, διευρυμένης ευρυζωνικής σύνδεσης για κυρίως για τους πολίτες που δεν ζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Φιγκυρέιντο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ κρίνω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση. Ξέρουμε ε, πόσο μεγάλη σημασία έχει η έννοια της καθολικής υπηρεσίας και πόσο το αριθμός 112 θα πρέπει να είναι γνωστό στη σπάση. Ε, κάτω από 30% των πολιτών γνωρίζουν αυτή τη στιγμή την ύπαρξη αυτού του αριθμού 112. Καταδεικνύεται ως εκ τούτου η ανάγκη συνέχισης των εκστρατιών ενημέρωσης και της διαμόρφωσης όλων των μέσων του ραδιοφώνου, του διαδικτύου, των ευηζωνικών συνδέσεων, ε, αλλά εγώ θα ήθελα να επιμείνω σε κάτι άλλο. κρύο τον κόδινο του κινδύνου. Ας μην χρησιμοποιηθεί αυτό για να ενισχυθεί η ε, κοινωνική αποξένωση.

Ε, γύρω στα 100 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν γύρω από το όριο της φτώχειας ε, με προφανείς δυσκολίες ε, πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες άρα θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμένες δράσεις για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση για όλους ανεξαρτήτως προϋποθέσεων. Δηλαδή κάποιος που δεν έχει λεφτά για να το πω απλά θα πρέπει να έχει παρόλα αυτά σύνδεση στις νέες τεχνολογίες και παρόλα αυτά σύνδεση στην καθολική υπηρεσία και κυρίως τον αριθμό κλίση έκτακτης ανάγκης 112. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, υποστηρίζω την έκθεση αυτή της κυρίας Ράπτη σχετικά με την καθολική υπηρεσία και τον αριθμό κλήσης έκτακτη ανάγκη 112. Πρέπει να προσπαθήσουμε αυτή η υπηρεσία να γίνει προσβάσιμη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και περισσότερο αποτελεσματική και θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού του σημείου από το οποίο ξεκινά η κλίση, ούτω ώστε να μπορούν να παρασχεθούν ιατρικές βοήθειε στον καλούνται αν αυτό είναι απαραίτητο Επίσης θα πρέπει να αποφύγουμε την ασφαλμένη χρήση ε, αυτού του αριθμού για φάρσες ε, ή ε, με άλλες μορφές κατάχρησης αυτής της υπηρεσίας. Δεν θα πρέπει τη στιγμή που κάποιος χρειάζεται αυτόν τον αριθμό έκτακτη ανάγκη, κάποιος άλλος να χρησιμοποιεί αυτόν τον αριθμό για να μπορεί να διασπείρει ασφαλμένα μηνύματα. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία σε πολλές γλώσσες, διότι κινούνται οι πολίτες της Ευρώπης σε όλες τις χώρες ε, και δεν μπορούν πάντοτε να μιλούν τη γλώσσα της κάθε χώρας. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμες, λοιπόν οι γλώσσες, οι πιο κοινέ γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία αυτή. Επίση, θέλω να τονίσω και τη σημασία της ε, προσβασιμότητας σε ιατρική βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Σκέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για τους πολίτες της Ευρώπης. Γι' αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια για το θέμα αυτό. Πολύ συχνά το σημαντικό έργο που γίνεται δεν φτάνει μέχρι τους πολίτες. Η δημοσιότητα πολύ συχνά στα κάτι μελη είναι αρνητική δημοσιότητα, αλλά τα θετικά σημεία σπανίως φτάνουν στη δημοσιότητα μόνο 26% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωρίζουν σχετικά με την ύπαρξη αυτού του αριθμού έκτακτης ανάγκης και γι' αυτό θα έπρεπε να θέσουμε το ερώτημα γιατί δεν είναι γνωστό και ποιος ευθύνεται για το ότι δεν είναι γνωστός αυτός ο αριθμός. Ε, υπάρχει ε, όλη η κατηγορία των πολιτών με ειδικέ ανάγκες αλλά και οι απλοί πολίτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον αριθμό και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να φτάσει το μήνυμα για τον αριθμό αυτό σε όλους τους πολίτες για να μπορούν να δουν και τη θετική θετική εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι λυπηρό ότι την αγνοούν ε, οι πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Θα ζητήσω από την Επίτροπο Μάλστρομ να μας πει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτό τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ. Η Επιτροπή πιστεύει ότι είναι εξαιρετική προσπάθεια και θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγητή την κυρία Ράπτη για τη δουλειά που έχει κάνει όπως επίσης και τις Επιτροπές ΙΝΚΟ ε, και για την έκθεση αυτή και πάλι. Όσον αφορά την Καθολική Υπηρεσία, χαίρομαι γιατί η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο βρίσκονται ε, στην ίδια πλευρά όταν μιλάμε για το ρόλο τον οποίο μπορεί να παίξει η Καθολική Υπηρεσία στον τομέα της ευρυζωνικότητας. Είναι ένα δίκτυο ασφαλείας που μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν θα εμποδίζονται οι πολίτες στο να συμμετέχουν ε, λόγω της έλλειψης επαρκών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η Καθολική Υπηρεσία δεν είναι μόνο τρόπο για να επιτύχουμε την ευρυζωνικότητα και θα πρέπει να έχει τη σωστή τη θέση μέσα στο οπλοστάσιο των μέτρων που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι νομικές υποχρεώσεις δεν θα επιβαρύνουν άδικα τις, τηλεπικοινων... τηλεπικοινωνιών, ούτε θα αυξάνουν άδικα τις τιμές προς τους καταναλωτές. Θα πρέπει η ευελιξία να ασκηθεί με τρόπο συνεκτικό και συνεπή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση επιτόπου και λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στη βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών, στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και στους πολίτες. Έχει αναφερθεί η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την Καθολική Υπηρεσία σε ένα ευρυζωνικό περιβάλλον μετά από τις διαβουλεύσεις πέρυσι. Θέλουμε να δείξουμε την προθυμία μας να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη στη διαδικασία εφαρμογής, δίνοντας κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή ε, των ε, υφισταμένων υπηρεσιών, καθολικών υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στην έκθεση συζητάμε με τα κράτη-μέλη για το περιεχόμενο των, μετρών, των μέτρων αυτών ε, και ε, θα δοθούν οι κατάλληλε γνωμοδοτήσεις σύντομα. Ο ρόλος του αριθμού 112 θεωρούμε ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο, ε, ότι είναι σημαντικός και θα πρέπει να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την πρόσβαση στον αριθμό 112 για άτομα με ειδικέ ανάγκε. ειδικές ανάγκες θα πρέπει να προωθήσουμε και τον εντοπισμό του τόπου από τον οποίο γίνεται η κλίση. Χρειάζεται πρόοδο στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και πιστεύουμε ότι θα είναι μια σωστή προσέγγιση για να βελτιώσουμε τα κοινά στάνταρτ αποδόσεων. Η Επιτροπή πιστεύει ότι ο αριθμός 112 θα είναι αποτελεσματικός εφόσον έχουμε ενημερώσει τους πολίτες για την ύπαρξη του αριθμού 112 για να γνωρίζουν ότι είναι ένας αριθμός που τους προστατεύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειες προώθησης του 112. Βασιζόμαστε και στη συνεργασία των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προωθήσει την ανταλλαγή πρακτικών και βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά ε, τα θέματα αυτά, ιδίως με την αναθεώρηση των κανόνων για το 112 και με την ε, προτυποποίηση και σας διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσει η Επιτροπή να συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε υψηλή απόδοση των ε, συστημάτων του αριθμού 112 με τρόπο συμβατό λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τεχνολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Η συζήτηση για τον αριθμό κλίση έκτατης ανάγκης 112 ολοκληρώθηκε εδώ. Και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα που είναι η έκθεση της κυρίας Άννα Μαρία Κοράτσα Μπίλτ για μια πιο αποτελεσματική και πιο